Καλημέρα. Ξεκινούμε τη συνεδρίασή μας. Πρώτο θέμα, έγκριση της σημερινής διάταξης. Αν δεν υπάρχουν προτάσεις για αλλαγέ. εγκρίνεται. Δεύτερο σημείο, έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων που έγιναν στις 30 Μαΐου και στις 8 Ιουνίου. Αν δεν υπάρχουν σχόλια, εγκρίνονται. Τρίτο σημείο. Ανακοινώσεις Προέδρου. 3.1. Επίσκεψη Καταρίνα Μασελίνου, Πορτογαλίδας Υπουργού, για ζητήματα ηθαγένειας και ισότητας. Είχε προγραμματιστεί να γίνει η επίσκεψη αυτή στη σημερινή μας συνεδρίαση, ωστόσο δυστυχώς η Γραμματεία ε, ενημερώθηκε ότι δεν μπορεί να παραστεί σήμερα η κυρία Μαρσελίνο και θα ε, αναβληθεί για κάποιο σημείο στο μέλλον η επίσκεψη, επίσκεψη αυτή. 3-2. Μέσω γραπτής διαδικασίας 23 και 28 Ιουνίου οι συντονιστές της Επιτροπής μας αποφάσισαν να συνταχθεί έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για την κατάσταση των γυναικών με αναπηρίες και να ανατεθεί στο ΕΛΚ για δύο πόντους να συνταχθεί έκθεση ιδιαίτερη πρωτοβουλία για μια στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του καρκίνου των γυναικών και να ανατεθεί στο EFDD, πάλι για δύο βαθμού πόντου, να συνταχθεί σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με τις ενωσιακέ προτεραιότητες εν ώψη της επερχόμενης συνόδου UNCSW 62, να αναβληθεί η αποστολή στην Σουηδία που είχε προγραμματιστεί για το Δεκέμβριο 2017 και να πάει στην επόμενη χρονιά και να ακυρωθεί η συνεδρίαση της 31ης Αυγούστου της Επιτροπής μας και να ψηφίσουμε σήμερα, σήμερα για τις ε, τροπολογίες στον προϋπολογισμό δίνοντας ε, και στην, στον εισηγητή μας την εντολή προκειμένου να κάνει τις σχετικές αλλαγές ε, με, στη θέση του Συμβουλίου. Αυτά. Λοιπόν, επόμενο θέμα είναι Προεδρία Συμβουλίου και παρουσίαση του προγράμματος αυτής από τον ε, Γευγένιο Σινόφσκι, που είναι Υπουργός Υγείας και Εργασίας της Δημοκρατίας της Εσθονίας. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω εδώ στην Επιτροπή σας για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα που είναι τμήμα του χαρτοφυλακίου μου ως Υπουργού. Είναι όμως πολύ σημαντική προτεραιότητα. Θα ήθελα, καταρχάς, να μιλήσω για την σημασία της ισότητας των φίλων. Το έχω ξαναπεί αυτό. Ε, η ανισότητα είναι απάνθρωπη, γιατί η ανισότητα είναι πάντα πείμα της διάκρισης και δεν θεωρεί ένα άτομο άτομο. Ε, η άνηση μεταχείριση είναι επίσης ηλίθια, χαζή, γιατί δεν είναι ρεαλιστική. Δεν χρησιμοποιούμε το δυναμικό που έχει ο άνθρωπος, ε, εφόσον οι γυναίκες δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες. Είναι επίσης ε, ε, και επικίνδυνο, γιατί Επίσης, ε, δημιουργεί κατακαιρματισμό στην αγορά εργασίας, οικονομική εξάρτηση και άνηση, άνισο βάρος, ας πούμε. Ε, επίσης, είναι βασικό αίτιο βίας και προφανώς οι γυναίκες αισθάνονται τη βία και έχουν αυτή την εμπειρία παντού σε όλο τον κόσμο. Για αυτούς τους λόγους λοιπόν ε, το να προωθήσουμε την ισότητα των φύλων ε, πρέπει να είναι βασικό στόχος στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ισότητα των φύλων δεν είναι μόνο ηθικό θέμα, είναι, βρίσκεται στην καρδιά της δημοκρατίας. Τα, όταν οι γυναίκες και τα παιδιά αντιμετωπίζουν τις ίδιες, ε, έχουν τις ίδιες ευκαιρίες, τις αντιμετωπίζουν με το ίδιο, αυτό οδηγεί σε πολιτική και οικονομική πρόοδο. Επομένως, ε, με μεγάλη χαρά μπορώ να σας πω ότι μου αρέσει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισφέρει πολύ σε αυτό το επίπεδο. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάει πάντα για την ε, ισότητα των φύλων και μιλούσε από τη δημιουργία της. Η ισότητα των φύλων για μας είναι προϋπόθεση για την ένταξη μιας χώρας και η χρηματοδότηση των προϋποθέσεων καθώς και η υποβολή τέτοιων στοιχείων στην εξωτερική πολιτική πάντα μπαίνει συζητήσει με τι τρίτε χώρε. Μην ξεχνάτε ότι πουθενά αλλού στον κόσμο δεν έχει επενδύσει και δεν έχει επιτύχει τόσα πολλά στην ισότητα των φύλων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι ικανοποιημένο που του επόμενου 6 μήνε η Εστονία μπορεί να συνεισφέρει στι πρωτοβουλίε Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα αυτό. Καταρχά, είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε ακόμα ένα βήμα για να αναπτύξουμε τις προϋποθέσεις, ούτως ώστε να εξορροπήσουμε την εργασία και την οικογενειακή ζωή. Ε, μέτρα τα οποία θα υποστηρίξουν ε, τον ίσο καταμερισμό των βαρών ανάμεσα στους γονείς είναι πολύ σημαντικά για να δώσουν στις γυναίκες την ε, δυνατότητα να συμμετέχουν περισσότερο στην ε, αγορά εργασία και στους άντρες την δυνατότητα να συνεισφέρουν περισσότερο στην οικογενειακή ζωή. Στην Αστωνική Προεδρία θα εστιάσουμε στις πρώτες συζητήσεις για το φιλόδοξο σχέδιο οδηγίας για την ισορροπία οικογενειακής ε, ζωής και εργασίας. Ε, θα, γίνουμε, θα γίνουν πολύ συγκεκριμένα βήματα για αυτή την εξισορρόπηση στην ε, συζήτηση που θα γίνει στην άτυπη υπουργική ε, στο Τάλιν ε, τον Ιούλιο των Υπουργών Εργασίας, ε, συγγνώμη, Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικογένειας και Ισότητας των Φύλων. Ε, σε αυτή την άτυπη θα επικεντρωθούμε στην ισορροπία ε, εργασίας ε, και οικογενειακής ζωής ε, στα πλαίσια των νέων μορφών εργασίας και οικογένειας. Ε, εμείς έχουμε μεγάλο χάσμα στην Εστονία ανάμεσα στους μισθούς ανδρών και γυναικών και αυτό μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε τα προβλήματα της, του διαχωρισμού στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο της πλατφόρμας του, του Πεκίνου ε, και τις σχετικές δράσεις θέλουμε να υιοθετήσουμε συμπεράσματα του Συμβουλίου ε, για αυτό το θέμα. Ε, επίσης, θα ξεκινήσουμε τον Οκτώβριο στις 11 στις Βρυξέλλες με μια εκδήλωση, η τρίτη εκδήλωση για τον δίκτυ ισότητας ανδρών και γυναικών. περίπου 300 άτομα θα συζητήσουν τα απορίσματα από τον δίκτυ για την ισότητα των φύλων. Ε, σε ό,τι αφορά τον επιμερισμό των βαρών και την οικονομική εξάρτηση των γυναικών, η κάθετη, ο κάθετος διαχωρισμός είναι τεράστιο θέμα. Ε, πολύ λίγες γυναίκες φτάνουν στα, σε ανώτατα κλιμάκια, στον ιδιωτικό τομέα, ε, στην, στα πανεπιστήμια, στην επιστήμη, στην τεχνολογία κτλ. Για να μην μιλήσω για την κυβέρνηση και την πολιτική. Η κυβέρνηση, η Κομισιόν έχει προτείνει ένα σχέδιο οδηγία για την ισότητα των φύλων ε, στα δουσού των εταιριών και λύσεις για να ρυθμιστεί αυτό το πρόβλημα. Τα κράτη-μέλη προσεγγίζουν διαφορετικά αυτό το πρόβλημα. Το Συμβούλιο προσπαθεί να φτιάξει ένα κείμενο αρκετά ευέλικτο. Στι συζητήσει επί Μαλτέζικη Προεδρία ε, προέκυψε ξεκάθαρα ότι πολλά κράτη-μέλη θα θέσουν το θέμα τη επικουρικότητα. Αν αλλάξει η κατάσταση των κρατών μελών, θα σκεφτούμε του καλύτερου τρόπου για να προωθήσουμε την πρόταση αυτή. Το 2017 θεωρείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως η χρονιά καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών. Πιστεύουμε ότι η βία κατά των γυναικών πολύ συχνά θεωρείται ιδιωτική υπόθεση και επομένως ε, υποτιμούμε τη σημασία της. Το γεγονός ότι διαπρόνται αυτά τα εγκλήματα από τους ε, συγγενείς των γυναικών θα πρέπει να είναι επιβαρυντικό στοιχείο και όχι ελευθερικό στοιχείο. Η ισότητα των φύλων είναι βασική αξία και θα πρέπει να ισχύει και να φαίνεται στην νομοθεσία, στην πρακτική, στην ομολογία και στην καθημερινή ζωή. Θα ήθελα να σα ενημερώσω για τι τελευταίε εξελίξει για τη διαδικασία επικύρωση τη σύμβαση τη ε, Κωνσταντινούπολη στην Εστονία. Το νομοσχέδιο τη ε, επικύρωση έχει περάσει από την πρώτη φάση στο Κοινοβούλιο και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο. Η ένταξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στην σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα σε όλο τον κόσμο και κατά τη διάρκεια τη Μαλτέζικη Προεδρία, το Συμβούλιο υιοθέτησε αποφάσει για την υπογραφή τη σύμβαση. Υπογράφτηκε εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση στι 13 Ιουνίου του 2017 και είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δυναμική. Το δεύτερο τμήμα του πακέτου που προτάθηκε από την Κομισιόν, η απόφαση για την ολοκλήρωση ε, και είμαστε έτοιμοι για να σημειώσουμε πρόοδο. Ε, θα συζητήσουμε καταρχά του ιστορικού κανόνε υπό τη μορφή ενό κώδικα διοντολογία. Αυτό θα θέσει τα θεμέλια για το πώ θα συμπεριφερθούν τα κράτη-μέλη και τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την εφαρμογή τη σύμβαση. Ε, είναι παράδοση ανάμεσα στο Τρίτο των Προεδριών και το πώ κινούμαστε, το πώ λειτουργούμε και ακριβώ μέσα αυτή την παράδοση θα υπογράψουμε την κοινή δήλωση του τρίου για την ισότητα των φύλων μαζί με τη Βουλγαρία και την Αυστρία. Στη δήλωση αυτή θα μιλήσουμε για τι προτεραιότητε των προεδρίων του τρίου του επόμενου 18 μήνε. Τελευταίο στοιχείο. Ε, θα ήθελα να σα μιλήσω για την ε, χάρτα, για την ποικιλομορφία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και το ετήσιο φόρουμ που γίνεται με όνομα ε, ποικιλομορφία και ηγετικό ρόλο στον κόσμο του ε, που θα γίνει στο Τάλιν τον Νοέμβριο 6 και 7, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, είναι μια ειδική εκδήλωση, ε, το πρώτο φόρουμ για την πρόθεση της ποικιλομορφία ε, στην Ανατολική Ευρώπη και οργανώνεται ούτως ώστε να ανταλλάξουμε καλές πρακτικές και να μιλήσουμε για το πώ προωθείται η ισότητα των φύλων σε διάφορε οργανώσει. Έχει κάνει πάρα πολλά η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα. Ε, η ισότητα των φύλων ε, δεν, ε, δεν σημαίνει ότι ό,τι κερδίζει ο ένας το χάνει ο άλλος. Σε καμία περίπτωση. Είναι μία μάχη, ε, αλλά δεν είναι μία μάχη μεταξύ των φίλων. Είναι μία μάχη για την ισότητα. Παρότι η πρόοδος είναι αργή, εγώ έχω πολλές ελπίδες και μπορώ να σε επιβεβαιώσω ότι έχουμε, είμαστε αποφασισμένοι να φέρουμε πιο κοντά την Ευρώπη σε μια ίση κοινωνία όπου όλοι θα αξιοποιούνται. Σας ευχαριστώ Υπουργέ. Για τις ε, ε, για την παρουσίαση του προγράμματος της Θεσσαλονικής Προεδρίας. Ο λόγος στα μέλη μας. Πρώτα ο λόγος ε, στους συντονιστές. Η κυρία Κασβάφα Βιέρε. Ξεκινά. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό για τα πολύ αισιόδοξα λόγια που μας είπε όσον αφορά το πρόγραμμα ε, εργασιών της ε, Εστονικής Προεδρίας αλλά και όσον αφορά τις αντιλήψεις της εστονικής κυβέρνησης σχετικά με την ισότητα των φίλων, όπως μας τις παρουσίασε. Διότι τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο και αυτονόητο σε συνθήκες και σε διάφορα νομικά έγγραφα βεβαίως έχει κατοχυρωθεί η ισότητα των φύλων, ωστόσο στην πράξη σε πολλούς τομείς ε, έχουμε μείνει πίσω. Γι' αυτό και το σκεπτικό που μας παρουσιάσατε νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε ορισμένες διαστάσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε σχετικά με τη σχέση οικονομίας και ισότητας. Πολύ συχνά η ισότητα ε, γίνεται κατανοητή ως μια μορφή δικαιοσύνης. Ε, ακριβώς επειδή θεωρούμε ότι αυτό το γυάλινο ταβάνι που ε, αναφέρουμε πολύ συχνά για τις γυναίκες είναι άδικο, ε, θεωρούμε ότι ως αδικία πρέπει να καταπολεμηθεί. Όμως υπάρχουν και πολύ ευρύτερα επιχειρήματα υπέρ της ισότητας που εδράζονται στην οικονομία. Η, διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι μια σπατάλη από οικονομικής σκοπιάς. Σκαπα, σπατάλη δυνατοτήτων και πόρων. Είναι και αυτό σημαντικό να φωτιστεί, διότι υπάρχουν μια σειρά από μέτρα και μια σειρά από τομείς που μπορούν να οδηγήσουν στο στόχο της πλήρους ισότητας. Και νομίζω ότι αυτή η κατεύθυνση είναι πολύ σημαντική και χαίρομαι που την ε, συμμερίζεται και η Εστονική Προεδρία. Βεβαίως ε, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν προβλήματα στο Συμβούλιο. Πολλοί επικαλούνται την αρχή της επικουρικότητας Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλιστεί βεβαίως ότι ε, ό,τι γίνει θα γίνει εντός των αρμοδιοτήτων που έχουν εκχωρηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η νέα λύση λοιπόν προτείνει συγκεκριμένα μέτρα ε, σε μια σειρά τομεί. Παρ' όλα αυτά θα παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον τις συζητήσεις και θα σας υποστηρίξουμε όπου χρειαστεί. Για την ε, Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Η σύμβαση αυτή έχει ε, υπογραφεί μένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εν μέρη μόνο ως προς τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκεκριμένα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω σκοπεύετε να ξεκινήσετε τη διαδικασία για την ε, υιοθέτηση και ευρύτερων συμφωνιών για την πλήρη και απόλυτη εφαρμογή της σύμβασης αυτής στα κράτη-μέλη. Διότι ε, η υπογραφή από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι μερική και μόνο. Ακριβώς γιατί περιορίζεται στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφορά το άσυλο, την ε, παράνομη διακίνηση ανθρώπων, αλλά όχι όλους τους τομείς της ζωής. Όπως και να έχει, θα ήθελα να εκφράσω το θαυμασμό μου για τον συστηματικό τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεται τα ζητήματα ε, στο πλαίσιο της Προεδρίας σας την ψηφιοποίηση, την οποία βεβαίως δεν αναφέρατε, ε, ξέρουμε ότι είστε ηγέτες σε, σε αυτό τον τομέα στον κόσμο ε, και νομίζω ότι και από αυτή την άποψη έχει να προσφέρει η ψηφιοποίηση κάτι στην ισότητα των φίλων. Ευχαριστώ κύριε Πέρας. Ευχαριστώ. Καταρχάς θα ήθελα προφανώς καταρχήν να ευχαριστήσω τον Υπουργό, ο εμφανίστηκε εδώ στην Επιτροπή μας. Όπου μιλάμε, προσπαθούμε να προωθήσουμε πρωτοβουλίες για την ισότητα των φύλων. Για να καταπολεμήσουμε την ανισότητα, να φτιάξουμε μια κοινωνία πιο ίση, πιο δίκαιη. Ε, σε ό,τι αφορά τις γενικές αρχές που ανέφερε, προφανώς συμφωνώ. Αυτός πρέπει να είναι ο, στόχος μας, ο στόχος μας και ακριβώς επ' αυτών των θεμάτων θα πρέπει να προσπαθήσουν τα διάφορα θεσμικά όργανα για να υλοποιήσουν αυτούς τους στόχους. Αυτό που λείπει, αυτό που είναι σημαντικό και όλοι πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει και πολιτική βούληση για να υλοποιήσουμε όλες αυτές τις μεγάλες, υψηλέ γενικές αρχές. Ε, και τώρα που εσείς ξεκινάτε την Προεδρία σας, ελπίζουμε να δώσετε αυτό το περιθώριο της εμπιστοσύνη, αυτή την όθηση, αυτή τη δυναμική. Πιστεύω ότι θα κάνετε τη διαφορά για να υπάρξουν σημαντικές πρωτοβουλίες για την ισότητα των φύλων. Αλλά δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι περάσαμε αυτή τη θητεία ε, ακούγοντας μεγάλες και υψηπετείς αναγγελίες για την ισότητα των φύλων και τίποτα δεν έγινε. Οι γενικές αρχές στις οποίες αναφερθήκατε μπορούν να υλοποιηθούν όμως με συγκεκριμένες πολιτικές. Καταρχάς, να υπογράψουμε τη σύμβαση της ε, Κωνσταντινούπολης. Χαίρομαι που θα η χώρα σας θα υπογράψει το Σεπτέμβριο του 2017 τη σύμβαση αυτή είναι η τελική τζίφρα, η τελική υπογραφή. Νομίζω ότι όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν επαρκή χρόνο για να μελετήσουν την επίπτωση που θα έχει αυτή η επικύρωση και νομίζω ότι καλό είναι να κάνουμε όλοι αυτό το βήμα. Είναι σημαντικό να υπάρξει αυτή η ευρωπαϊκή επικύρωση για να υλοποιήσουμε τη δέσμευση. Και μαζί με την Επιτροπή Ελευθεριών ε, υποβάλαμε μία έκθεση της ε, του Κοινοβουλίου ε, για αυτή την σύμβαση της Κωνσταντινούπολη, ούτως ώστε να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσει ε, των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων ε, στα πλαίσια της καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών. Τώρα, για την συμφιλίωση οικογενειακής ζωής και εργασίας. Άκουσα τον συνάδελφο από το, από το ΕΛΚ να μιλάει για αυτό το θέμα. Νομίζω ότι μιλήσατε για, για οδηγία για την άδεια, για τις άδειες καλοκαίρι, για τις διακοπές, εν Αυτό άκουσα από την Ισπανική καμπίνα. Δεν ξέρω αν ήταν αυτό. Πώς νομίζετε, πώς νομίζετε ότι θα συμβιώσουμε την οικογενειακή ζωή με την ε, εργασιακή ζωή. Το θέμα δεν είναι να πάρουμε διακοπές. Όχι, δεν συμφιλιώνουμε έτσι αυτά τα δύο κομμάτια της ζωής μας, παίρνοντας διακοπές. Το θέμα είναι να, μπορέ, να μπορούμε να μπορούμε να παίρνουμε άδεια, γονική άδεια, ούτω ώστε να μπορούμε να συμφιλιώσουμε αυτά τα δύο κομμάτια της ζωής. Και η γονική άδεια δεν είναι διακοπές, καλοκαιρινές ή άλλου τύπου, αυτό άκουσα λοιπόν. Προσοχή να μην μπερδεύουμε αυτά τα πράγματα. Η, οδηγία για τι διακοπέ είναι κάτι άλλο. Ελπίζουμε να κινηθεί γρήγορα το Κοινοβούλιο, να πάρει θέση γρήγορα και το Συμβούλιο να αισθανθεί την ανάγκη να διαπραγματευτεί μαζί μας. Επίσης, η οδηγία ε, για την μητρότητα, ε, επειδή δεν υπήρχε συμφωνία στο Συμβούλιο χρειάστηκε η Επιτροπή να, το, να την αποσύρει. Επίσης, η οδηγία για τις γυναίκες στα Δουσού. Εάν εμείς που είμαστε εδώ πέρα, σε αυτό το κοινοβούλιο, όπου εδρεύουν τόσε πολλέ διαφορετικέ ε, απόψεις, κόμματα κτλ. Καταφέρνουμε να τα βρίσκουμε παρόλα αυτά και μετά ε, τρώμε στα μούτρα την πόρτα του Συμβουλίου, ε, είναι κρίμα. Νομίζω δεν έχει νόημα έτσι. Εμείς μιλάμε και τελικά δεν βγαίνει τίποτα. Πρέπει να αναλάβουμε όλοι μας την ευθύνη, όχι μόνο ένα κράτος μέλος, όχι μόνο η χώρα της Προεδρίας κάθε φορά. Πάντως, στην Προεδρία θέλω να πω αυτή τη στιγμή να κάνει μια προσπάθεια, ούτω ώστε να προκαλέσει το ενδιαφέρον στο εσωτερικό του Συμβουλίου, τουλάχιστον για να γίνει μια διαπραγμάτευση. Αυτή τη στιγμή στο Κοινοβούλιο έλαβε θέση. Αυτά και σας ευχαριστώ ακόμα μια φορά για την ε, παρουσία σας σε αυτή την Επιτροπή. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία, γιατί οι δικές σας επιτυχίες θα είναι και δικές μας. Θα είναι επιτυχίες όλων των ανδρών και γυναικών που πιστεύουν σε μια πιο δίκαιη ευρωπαϊκή κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ. Να σας ευχαριστήσω και εγώ εκ μέρους των φιλελευθέρων, κύριε Υπουργέ, για την παρουσία σας εδώ και για την παρουσίαση που κάνατε. Θέλω να συμφωνήσω με τη συνάδελφα από τους σοσιαλιστές. Χρησιμοποιήθηκε όρος δυσαρέσκεια από εσάς. Πράγματι, είμαστε δυσαρεστημένοι εμείς που κάνουμε αυτόν τον αγώνα για την ισότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα τον εγκαταλείψουμε. Σας ευχαριστούμε για το γεγονό ότι μας ενημερώσατε για την ε, κύρωση από πλευρά της Εστονίας της Σύμβασης Κωνσταντινούπολης. Είναι πολύ θετικό αυτό. Σχετικά με την, ε, με την ένταξη του, των θεμάτων ισότητας ε, στο θεματολόγιο για την ψηφιοποίηση. Ε, θα ήθελα, όπως είπε και η συνάδελφος από το ΕΛΚ, θα ήθελα να σας ρωτήσω, μιας και είστε ηγέτες σε αυτό το τομέα, σε παγκόσμιο επίπεδο, ε, έχετε μήπως ιδέες για το πώς, να μπορούμε να εντάξουμε τις γυναίκες στο ψηφιακό θεματολόγιο και τα ζητήματα της ισότητας. Όσον αφορά τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια, θέση που εκφράσατε ήταν να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όταν περιμένουμε απλά να δούμε, σε οποιοδήποτε τομέα που άπτεται των ε, ίσων δικαιωμάτων, δεν πρόκειται να επιτύχουμε τίποτα. Θα ήθελα λοιπόν να σας καλέσω να αναλάβετε πρωτοβουλίες και συγκεκριμένες ε, κινήσεις προς την κατεύθυνση της επίτευξης της ισότητας των δύο φίλων. Η κυρία Βαλίνα. Ε, ευχαριστώ. Καλημέρα. Καταρχάς πρέπει να σας ευχαριστήσω Υπουργέ για την παρουσία σας που ήρθατε εδώ για να μας εξηγήσετε τις προτεραιότητες στον τομέα το δικό μας. φαντάζομαι ότι τα φαινόμενα ανισότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μας δημιουργούν προβλήματα και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων ε, βλέπουμε ότι η ανισότητα είναι στο ύψος του 52,9% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, έχουμε τρία χρόνια μέχρι το 2020 και είπατε κι εσείς ότι χωρίς πραγματική πολιτική βούληση, χωρίς μέτρα αποτελεσματικά για να προωθήσουμε την ισότητα, μόνο με λόγια δεν πρόκειται να υλοποιηθούν οι στόχοι για την, για την ισότητα που έθεσε η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση τον εαυτό της για αυτή τη χρονιά στα πλαίσια της στρατηγικής για την ισότητα. Να μην ξεχνάμε το γεγονός ότι έχουν υπαναχωρήσει τα δικαιώματα των γυναικών ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολλές χώρες, όπως τη δική μου Φερρυπίν. Λαμβάνοντας υπόψη ε, την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, θέλουμε 70 χρόνια να φτάσουμε σε ισότητα. 40% για να υπάρξει ε, πραγματική ε, ισότητα στο σπίτι. Ε, επίσης, 30 ε, χρόνια για να έχουμε ίσο μισθό και 20 χρόνια για να φτάσουμε σε ίση πολιτική εκπροσώπηση. Ε, προχωράμε, όπως είπατε και εσείς, αλλά αργά, πολύ αργά. Επίσης, επίσης είσαστε υπουργό Υγείας και Εργασίας στη χώρα σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν τι μέτρα θα υιοθετηθούν κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας για να μειωθούν αυτά τα χάσματα ανάμεσα στα δύο φύλλα, αυτά τα κενά ιδίω στην εργασία και ειδικά στην οδηγία, σε ό,τι αφορά την οδηγία για τη συμφιλίωση μεταξύ εργασίας και οικογενειακής ζωής. Ένα άλλο σημαντικό θέμα στο οποίο αναφερθήκατε είναι η βία και φέτος το 2017 ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε ότι η χρονιά αυτή είναι η χρονιά όπου θα πρέπει να σταματήσει η βία κατά των γυναικών. Δυστυχώς όμως αυτό το, αυτή η μάστιγα της ε, βίας των ανδρών πλήττει όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη χώρα μου την Ισπανία και μέχρι στιγμής ε, το 2017 είχαμε 34 δολοφονημένες γυναίκες, αν και τα νούμερα ε, μερικές φορές μιλάνε για 59. 34, 34 γυναίκες που δολοφονήθηκαν από τους συντρόφους τους. Δηλαδή μιλάμε για ένα θύμα κάθε πέντε μέρες. Αυτή, όπως είπατε κι εσείς, η ανισότητα είναι μία από τις αιτίες της βίας αυτής. Επίσης, ε, αν κατάλαβα καλά, η χώρα σας μείωσε τη χρηματοδότηση των γυναικών που καταπολεμούν τη βία κατά των γυναικών με βάση τα όσα καταγγέλουν αυτοί που μας, ε, μας καταγγέλνουν διάφορες οργανώσεις της Εστονίας που ανήκουν στο τμήμα του Ευρωπαϊκού Λόμπι των Γυναικών ε, δεν μπορούν ε, λόγω των μειωμένων κονδυλίων να βοηθήσουν τα θύματα. Θα ήθελα να μας το σχολιάσετε αυτό. Χθε υιοθετήσαμε στην Επιτροπή μας μαζί με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών το ψήφισμά μας και ζητάμε μια πολύ γρήγορη επικύρωση της Σύμβασης της ε, Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και τη βία στο σπίτι. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε για ποια συγκεκριμένα μέτρα θα προωθήσει η Προεδρία σας, ούτως ώστε να προωθήσει μια διαδικασία επικύρωσης για όλα τα κρατημέλη. Όλα. Και να προωθήσει υπηρεσίες και στήριξη προς τα θύματα των, ε, της ε, βίας Τη ε, της βίας κατά των γυναικών και φυσικά εδώ μιλάμε και για τις ε, γυναίκες πρόσφυγες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Είναι πάντοτε πολύ θετικό το να έχουμε την ευκαιρία να συζητούμε τις προτεραιότητες της κάθε Προεδρίας, ιδίω στον τομέα της ισότητας των φαίνων. Ε, να ξεκινήσουμε με μια γενική παρατήρηση. Πολλοί από εμάς σε αυτή την Επιτροπή έχουμε την εντύπωση ότι η ατζέντα για την ισότητα των φίλων ε, έχει ε, πέσει σε δεύτερη μοίρα ε, και σε πολλούς τομείς έχει μπλοκαριστεί η πρόοδος. Θα ήθελα λοιπόν να σας καλέσω με την ευκαιρία της παρουσίας σας σήμερα εδώ να αλλάξετε τον ρου των εξελίξεων των τελευταίων ετών και να κινηθείτε σε μια διαφορετική κατεύθυνση. Νομίζω ότι έχετε όλε τις δυνατότητες να το κάνετε. Πέραν των ζητημάτων που αναφέρθηκαν ε, ήδη και της κατάστασης ε, των γυναικών στην Ευρώπη, όπου απέχουμε πάρα πολύ ακόμη από το να επιτύχουμε την πλήρη ισότητα των δύο φύλων. παρόλα αυτά, νομίζω ότι μπορείτε στη διάρκεια του εξαμήνου αυτού να κάνετε τρία πράγματα και θα σας βοηθήσουμε. Είπατε το θεματολόγιο ε, συνδυασμού προσωπικής επαγγελματικής ζωής. Εμείς είμαστε πολύ πιο φιλόδοξοι από το κείμενο της Κομισιόν, το οποίο πολλοί από εμά θεωρούμε ότι ε, είναι πραγματικά πάρα πολύ θέσει. Δηλαδή, πρώτον, περισσότερη φιλοδοξία σε σχέση με το κείμενο που μας παρουσίασε η Κομισιόν. Δεύτερον, η οδηγία για τη συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια που έχει μπλοκαριστεί αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο. Φυσικά δεν περιμένουμε η δική σας Προεδρία να ξεμπλοκάρει αυτό το πολύ δύσκολο φάκελο. Όμω, αν καταφέρουμε εντό του εξαμήνου τουλάχιστον να ξαναξεκινήσουν οι συζητήσει επί του θέματο αυτού, θα, θα, θα έκανε αυτό μια πραγματική διαφορά. Ε, και θα ξεκινούσε μια διαδικασία ε, που θα μπορούσε να οδηγήσει τουλάχιστον στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Αυτό είναι κάτι που μπορείτε να το επιτύχετε εντό του εξαμήνου. Και τρίτον, πρέπει να σα πω ότι το ήμουν πολύ χαρούμενο που το, το είδα και στο πρόγραμμά σα. Το ζήτημα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Βλέπω στι προτεραιότητέ σα ότι θέλετε να διευρύνετε το ρόλο του ΕΠΣΚΟ στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Αυτό είναι πολύ θετικό. Είναι ένα αίτημα ε, της Επιτροπής μας να λαμβάνονται υπόψη τα ζητήματα του φύλου στην ε, διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Αν λοιπόν μπορείτε να καταβάλλετε προσπάθειες και σε αυτή την κατεύθυνση, πραγματικά θα σας ήμασταν ευγνώμονες. Να ας σταματήσουμε να ανακόψουμε αυτήν την ε, τάση το ζήτημα της ισότητας των φύλων να μην αποτελεί και να μην θεωρείται γενικά ένα θέμα με στο οποίο πρέπει να επικεντρώνεται η Προεδρία. Ευχαριστώ, κυρία Αναγέτη. Eh, Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, για τα εισαγωγικά σας λόγια. Θα ήθελα να ξεκινήσω με αυτά που μόλις είπε ο προλαλής σας. 27 υπουργοί παρουσίασαν το πρόγραμμα της Προεδρίας τους για την ισότητα των φύλων. Χαίρομαι για τις μέχρι σήμερα επιτυχίες, μόνο που οι επιτυχίες αυτές έρχονται πολύ αργά. Αυτό με απογοητεύει πραγματικά. Με εξοργίζει, με εξαγριώνει. Ειδικά αν λάβουμε υπόψη μας τα προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας, με βάση την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περισσότερες αρμοδιότητες ε, για αυτά τα θέματα που αφορούν ε, την καθημερινότητα των ανθρώπων και που μπορούν να βελτιώσουν τόσο πολύ την κατάσταση των γυναικών. Και όμως η Κομισιόν και το Συμβούλιο δεν έκανε τίποτα ουσιαστικά. Βλέπετε πόσε γυναίκε είμαστε εδώ σήμερα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό και ενοχλητικό που τα πράγματα πηγαίνουν τόσο αργά στην Σουηδία, που είναι μια πολύ φεμινιστική χώρα. Βλέπουμε ότι ε, ακόμα και στη σύνταξη δεν είμαστε ίσοι. Δηλαδή, εμείς δεν είμαστε τόσο σημαντικές όσο οι άντρες, υπουργοί μου, κύριε Υπουργέ μου. Κοιτάξτε, εάν δεν γίνουν συγκεκριμένες προσπάθειες, δεν πρόκειται να πετύχουμε τίποτα, ούτε στο Συμβούλιο, ούτε αλλού. Παρ' όλα αυτά διατηρούμε την ελπίδα. Πρέπει να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο. Εσείς, Υπουργέ, μπορείτε να κάνετε όμως τη διαφορά. Αλλά πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προτεραιότητα σε αυτό το θέμα. Εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο κάνουμε ό,τι μπορούμε στην Επιτροπή μας. Και εσείς μπορείτε να κάνετε αυτό που είναι καλύτερο. Uh, Ευχαριστώ. Ε, ο λόγος στον Υπουργό για να μας απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ. Ε, πολλοί από εσάς εκφράσατε τη δυσαρέσκειά σας για την ανεπαρκή πρόοδο που έχει σημειωθεί. Συμφωνώ μαζί σας. Ούτε εγώ είμαι ευχαριστημένος. Δυστυχώς υπάρχουν ωστόσο κάποια όρια ε, στο τι μπορεί να κάνει μια Προεδρία μέσα σε 180 μέρα, ε, μέρες για ε, να διασκεδάσει αυτή τη δυσαρέσκεια. Θα κάνω ό,τι μπορώ όμως. Εν πάση περιπτώσει, ας ε, ε, απαντήσω λοιπόν στα συγκεκριμένα ζητήματα που τέθηκαν. Οδηγία για, την, για τον συμβιβασμό προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Το Συμβούλιο πολλές φορές έχει εκφράσει τη θέση του και την επιθυμία του να συνεχιστούν οι συζητήσεις πάνω στην πρόταση που έχει υποβληθεί και θέλουμε ήδη από την επόμενη εβδομάδα που θα γίνει η άτυπη συνάντηση ΕΦΣΚΟ να συζητηθεί αυτό το θέμα. Θα είναι ένα από τα βασικά θέματα που θα συζητηθούν, το, ζήτημα δηλαδή της, ε, του, ε, του συνδυασμού ε, και της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματική και προσωπικής ζωής. Είπατε ότι υπάρχει αυτό το ζήτημα της φιλοδοξίας. Ξέρετε πάντοτε, όποιο και αν είναι το πρόγραμμα μια προεδρία όταν παρουσιάζεται, άλλοι λένε ότι είναι πολύ φιλόδοξο, άλλοι λένε ότι είναι όχι αρκετά φιλόδοξο. Ε, όσον αφορά το ζήτημα τη ε, αναλογικότητα και τη επικουρικότητα και το ζήτημα των γονικών αδειών υπάρχει ήδη ισχύουσα νομοθεσία αυτό που θα κάνουμε εμεί ω Προεδρία είναι να καταγράψουμε τι απόψει των κρατών μελών και να προσπαθήσουμε να ε, βρούμε ένα συμβιβασμό. Πάντω, μέχρι στιγμή υπάρχουν ήδη δύο εθνικά κοινοβούλια τα οποία έχουν θέσει ζήτημα επικουρικότητα. Παρ' όλα αυτά, είναι σημαντικό το θέμα αυτό και προσβλέπουμε και στη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να προχωρήσουμε. Σύμβαση Κωνσταντινούπολη. Προφανώ χαιρετίζουμε την ενδιάμεση έκθεση που συνέταξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θεωρούμε ότι συμβάλλει θετικά και στις συζητήσεις που γίνονται στο Συμβούλιο. Πρόθεσή μας είναι να τηρούμε ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, για όλα τα θέματα και σε όλες τις φάσεις διαπραγμάτευσης, καθώς αυτή θα εξελίσσεται. Ενώ έχουν ήδη ε, συμφωνηθεί και στις συναντήσεις με τους ε, το φθινόπωρο. Ρωτήσατε για τη σχέση μεταξύ πληροφορικής και ισότητας των φύλων. Ξέρετε ότι υπάρχει ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου της πληροφορικής. Ωστόσο, δυστυχώς, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ψηφιακή λύση που θα μπορούσε να δοθεί στο ζήτημα το, της ισότητας των, των φύλων. Και προφανώς δεν μπορούμε να περιμένουμε από την πληροφορική να λύσει όλα τα προβλήματα ε, που ανακύπτουν. Ε, νομίζω ότι εδώ, σε αυτό το τομέα, οι πολιτικές στην παιδεία και στην απασχόληση θα είναι πολύ πιο σημαντικές προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Ε, υπάρχει βεβαίω και η πλατφόρμα του, του Πεκίνου που αναφέρθηκε για το ζήτημα της συμμετοχής γυναικών στα δυτικά συμβούλια. Προσωπικά συμμερίζομαι απόλυτα τη δυσαρέσκειά σας για την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα. Ωστόσο υπήρξαν χώρες οι οποίες ε, υπήρξαν χώρες ε, που στη διάρκεια της δικής τους προεδρίας κατέβαλαν προσπάθεια προκειμένου να ξεμπλοκαστεί το θέμα, χωρίς επιτυχία όμως. θα ήταν μη ρεαλιστικό να σας πω ότι θα σημειώσουμε πολύ μεγάλη πρόοδο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα το εγκαταλείψουμε βεβαίως. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι από την πλευρά μας θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας προκειμένου να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Κασλόφσκα θέλει να απαντήσει αν κατάλαβα σωστά. Ζητώ συγγνώμη, Πρόεδρε, που ξαναπαίρνω το λόγο. Θέλω να ξαναπάμε λίγο στο θέμα του ψηφιακού χάσματος. Είναι ένα νέο θέμα αυτό. Θα ήθελα να σας δώσω κάποια ενδιαφέροντα δεδομένα. Το θέμα δεν είναι ότι δεν υπάρχουν πολλές γυναίκες που δουλεύουν στον τομέα το ψηφιακό, ειδικά στα υψηλά κλιμάκια και στις διευθυντικές θέσεις. Το θέμα είναι ότι οι γυναίκες είναι πιο απίθανο να υποφεληθούν από τα ωφέλη του ψηφιακού κόσμου. Δεν χρησιμοποιούν δηλαδή τόσο πολύ ας τις ψωτικές τους κάρτες δεν πουλάνε πράγματα μέσω ίντερνετ ή δεν μαθαίνουν από το ίντερνετ. Εδώ έχουμε ένα χάσμα ύψους 15% το οποίο διευρύνεται με γοργό ρυθμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ξέρουμε ότι το μέλλον είναι ψηφιακό. Εμείς ε, στην Εστονία το ξέρουμε πολύ καλά. Επομένω, το ερώτημά μου είναι, υπάρχει περίπτωση κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας να μάθουμε περισσότερα για την κατάσταση που πραγματικά επικρατεί στα κράτη-μέλη και αν αυτά τα χάσματα ανάμεσα στα δύο φύλλα ε, διαφέρουν από κράτο σε κράτος. Γιατί εδώ μιλάμε για κάτι το οποίο είναι τεράστια σημασία. Και εμείς στην Εστονία ε, έχουμε την τάση να χρησιμοποιούμε πιο πολλές ψηφιακές λύσεις α, ε, περισσότερα από πουδήποτε άλλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, ίσως να έχετε περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα του χάσματος των δύο φύλων. Ο υπουργό για να αντιδράσει. Φυσικά. Ε, το χάσμα των φύλων ε, και σε επίπεδο δεξιοτήτων και γενικότερα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι δεξιότητες για την πληροφορική ειδικά είναι διαφορετικές από χώρα σε χώρα και οι γυναίκες εκπροσωπούνται τελείως διαφορετικά από τομέα σε τομέα και η, και η εκπροσώπησή τους ε, στο ψηφιακό κόσμο εξαρτάται από τις δεξιότητες που έχουν σε αυτό το επίπεδο. Εμείς ως χώρα έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ και σε επίπεδο εκπαίδευσης και στο δημόσιο τομέα και στην αγορά εργασία για να ενισχύσουμε τον κόσμο, να του δώσουμε τέτοιε δεξιότητε, ειδικά τους πιο ηλικιωμένου εργαζόμενου. Φυσικά θα μιλήσουμε στα συμπράσματα του Συμβουλίου για το χάσμα μεταξύ άντρων και γυναικών στο μισθό, ειδικά και ειδικά για το χάσμα αυτό που υπάρχει σε αυτούς που δουλεύουν στον ψηφιακό κόσμο, στον ψηφιακό χώρο. Άλλες ερωτήσεις? Σας ευχαριστούμε Υπουργέ που, που επισκεφθήκατε την ε, Επιτροπή μας και παρουσιάσατε τις ε, προτεραιότητές σας για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων. Σας ευχόμαστε σε προσωπικά και στην ομάδα σας καλή επιτυχία και θα περιμένουμε και αυτά τα απτά αποτελέσματα. Mm, Συνάδελφοι, επόμενο θέμα στη μέση διάταξη είναι Γενικός Προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, όλα τα τμήματα, εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης, η συγγήτρια, συντάκτρια δηλαδή της γνωμοδότησης, είναι η κυρία Μπάρμπαρα Ματέρα, αλλά εξ όσων γνωρίζω η κυρία Καζλόφς Χαραγέβιτς θα την ε, εκπροσωπήσει στη σημερινή συνεδρίαση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Μπάρμπαρα δυστυχώς δεν κατάφερε να έρθει σήμερα εδώ, παρόλα αυτά μου άφησε κάποιες σημειώσεις και θα σας τα διαβάσω. Τι θα σας τις διαβάσω. για να ακούσετε ποιες είναι οι σκέψεις της. Το 2018 η Επιτροπή ε, Γυναικών θα επικεντρωθεί στην εξασφάλιση χρηματοδότησης επαρκούς ε, για τα προγράμματα ε, ισότητας, ηθαγένειας την ε, διεύρυνση των, ε, της γυναικών σε, στον τομέα της πληροφορικής και αύξηση της παρουσίας ε, των γυναικών σε επιστημονικούς τομείς όπου υποεκπροσωπούνται. Αυτό έχει σημασία διότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο προϋπολογισμός ως αποτελεσματικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της ανισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να εξετάζονται και εν ώψη της προετοιμασίας του επόμενου πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου ε, συμπεριλαμβανομένης ε, μιας ε, δυνατότητας ορισμού κονδυλίων για την καταπολέμηση της ανισότητας ανδρών και γυναικών. Δύο ακόμα σημεία. Πρώτον, τα ενωσιακά προγράμματα και ταμεία όπως το ορίζοντας 2020 και τα ευρωπαϊκά κοινωνικά ταμεία θα πρέπει να υποστηρίζουν στεναρά τις γυναίκες στην επιχειρηματικότητα και ως προς την ε, πρόσβαση ε, σε χρηματοδότηση και τραπεζικά δάνεια. Επίσης, στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας των Φιλών θα πρέπει να δημιουργηθεί ε, μια ομάδα για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών προκειμένου να μπορούν να καταγράφονται στατιστικά στοιχεία και να λαμβάνονται μέτρα. Νομίζω ότι ε, είναι σημαντικό να ενταχθεί μια τέτοια λογική και στο ψήφισμα της Επιτροπής Προπολογισμού προκειμένου να επιτευχθούν οι αντίστοιχοι στόχοι και ελπίζω ο εισηγητής ο κ. Γιουρισσόν, θα λάβει υπόψη του τις δικές μας παρατηρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. No Comments. Άλλα σχόλια παρακαλώ. Πολύ ωραία. Και τώρα οι σκιώδεις εισηγητές. 25 Αυγούστου είναι η ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούμε να υποβάλουμε τροπολογίες. Αυτά. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Το επόμενο θέμα είναι οι ψηφοφορίες. Αλλά θα ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες στις 10.30. Σταματάμε μέχρι τις 10.30.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

And um, Συναδέλφοι, να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Έκτο σημείο της ημέρης σα διάταξη. Ενίσχυση των γυναικών, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναχέντ, έγκριση του σχεδίου έκθεσης, Να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Συμβαστική τροπολογία 9 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 79 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Στροπολογία 8, πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Για το δεύτερο τμήμα. Για τροπολογία 80, δεύτερο τμήμα. Ψηφίστε παρακαλώ, ένα ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρασε ψηφοφορία. It's rejected. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. MP2, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, όχι, Α, όχι, δεν ψηφίζεται το δεύτερο τμήμα. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, Τροπολογία 110. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Τροπολογία 110. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Καλύτερα να, το, ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Άρχισε τη ψηφοφορία. τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 112 πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, ξανά. Τροπολογία 112, δεύτερο, όχι, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Ωραία. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 112. 112 δεύτερο τμήμα. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Άρχισε η ψηφοφορία. Πέρασε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Εγκρίνεται, ωραία. Έμπλ 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 32 έμπλ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έμπλ 33 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έμπλ 34 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, 210 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 104 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 106 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 107 υπέρ, κατά, αποχές Απορρίπτεται. Τροπολογία 108 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έμπλ 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 113. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά καλύτερα. Ψηφίστε παρακαλώ. Άρχιτε ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Rejected. Απορρίπτεται. Amendment Τροπολογία 118 υπέρ, υπέρ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ηλεκτρονικά. Άρχισε η Για την τροπολογία 118. Ψηφίστε παρακαλώ τώρα. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 207 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 211 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 132 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έμπλη να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ωραία. Α ψηφίσουμε ηλεκτρονικά επί της συμβαστικής 15, παρακαλώ. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ε, έμπλ 3. Πρώτο τμήμα. Α, όχι. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 16. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά να το ελέγξουμε. Ωραία. Ας το ελέγξουμε λοιπόν. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 130 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ωραία, να το ελέγξουμε. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά τότε. Ψηφίζετε. Πέρσι προφορίες. Απορρίπτεται. Τροπολογία 131 υπέρ. Κατά. Αποχές. Καλύτερα να το δούμε. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρα στις προφορίες. Απορρίπτεται. Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 137 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έμπλη 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Τώρα. Πέρα στους ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. Από κοινού ψηφοφορία για, τις, ε, για την τροπολογία 141. Ε, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 144 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 173 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 175 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 184 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 187 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 191 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 193 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 146 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 147 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 148 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 149 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά τώρα. Πέρας προφορίας. Απορρίπτεται. 152 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 153 υπέρ. Κατά. εποχέ, Εγκρίνεται. 154 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 159 υπέρ κατά αποχές να το δούμε. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρασε ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 171 υπέρ, κατά, αποχές, να το δούμε. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά για να το ελέγξουμε. Πέρας προφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 172 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ωνα... Ε, ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά είπε, για την τροπολογία, τη συμβαστική τροπολογία 24. Πέραση τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Εκατόν τρία υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 204 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 205 υπέρ κατά, αποχές, να το δούμε, να το ελέγξουμε. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρας προφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 206 και έμπλη 35 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 26 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 94, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 28 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 29 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 30 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. ΕΜΠΙ 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. «192 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται». Συμβαστική 31 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έμπλη 37 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 178. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 179 υπέρ, κατά, αποχές. Να το ελέγξουμε. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά τώρα, πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2.19. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, να το δούμε, να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ τώρα της ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας, απορρίπτεται. Amendment 180 in favor. 180 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 181 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 182 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ας το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε για την 182. Πέρας προφορίας Απορρίπτεται. Έμπλ 18 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να το ελέγξουμε. Ψηφίστε παρακαλώ για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας αυτής. Πέρας προφορίας Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές. Να το δούμε. Ψηφίστε ηλεκτρονικά παρακαλώ τώρα. Άρχισε ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έμπλ ε, 19 ε, in favor. Έμπλ 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 189 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 197 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 138. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Παρακαλώ, ελέγχουμε ηλεκτρονικά για το πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω το ίδιο. Αλλά ας ελέγξουμε. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 142. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 143 υπέρ κατά αποχές ναι, ηλεκτρονικός έλεγχος ψηφίζουμε πέρασε απορρίπτεται 145 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 222 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται. Ε, τέλος. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, κατά πίπτη. Τροπολογία 223. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 224 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Εκτιμώντας ε, τροπολογία 16 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 32 υπέρ κατά αποχές έλεγχος ηλεκτρονικός άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Έμπλ α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές έγκρινεται. Έμπλ D υπέρ κατά αποχές έγκρινεται. Τροπολογία 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 25 υπέρ κατά αποχές τι λέτε. 25. Γιατί κρίναμε τη 41 και η άλλη είχε καταπέσει. Τροπολογία 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, ηλεκτρονικός έλεγχος. Τέλος. Απορρίπτεται. Έμπλ ε υπέρ κατά αποχές έλεγχος ηλεκτρονικός άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. F με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 ναι, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 31 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 34 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος ηλεκτρονικός άρχεται. The vote is closed. Adopted. I'm so sorry. It's my, mistake. Μάλιστα εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Amendment 62. Τροπολογία 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος ηλεκτρονικός πέρας απορρίπτεται 64 τώρα, η 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 65 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 69 υπέρ. Αποχές, έλεγχος ηλεκτρονικός, άρχεται. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6, υπέρ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Άρχεται. Τέλος. Απορρίπτεται. 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 58 υπέρ κατά αποχές έλεγχος παρακαλώ. Άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται.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 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 13, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 14, υπέρ, κατά, αποχές, α, απορρίπτεται. 15, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε. The vote is closed. It's adopted. Congratulations. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Πολύ καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε. Άννα, θέλεις το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τη συνεργασία όλους. Ήταν ε, σημαντικό ε, η έκθεση, η σημαντική έκθεση αυτή γιατί καλύπτει πολλά, πολλά, πολλές πτυχές. Ευχαριστώ λοιπόν όλους και όλος ιδιαίτερα στη Γραμματεία αλλά και τη Στεφανή και τον Έρικ που έκαναν εξαιρετική δουλειά. Ευχαριστώ και καλό καλοκαίρι σε όλους. Yeah, sorry. Yeah. Sorry. Now we are going to the uh, uh, second point on the agenda. Πάμε στο δεύτερο σημείο της ψηφοφορίας. Θεμελιώδη δικαιώματα, πτυχές μάλλον, ε, ε, θεμελιώδη δικαιώματα των Ρωμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά πολέμηση των ε, τσιγκάνων Τροπολογία 14, δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ. Against. Abstention adopted. Second part in favor. Against. Υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Check. Okay. Amendment 14, second part. The vote is open. Δεύτερο τμήμα. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Πέρας. Adopted. Amendment 15. First... Τροπολογία 15, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίπτεται. 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε ηλεκτρονικά τέλος εγκρίνεται 19 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 33 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται.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 αποχές εγκρίνεται. Εκτιμώντας τροπολογία 1 περ αποχές έλεγχος ηλεκτρονικός. Τροπολογία 1 για τα εκτιμώντας υπέρ κατά, ε, μάλλον άρχεται και τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ. Τροπολογία 2 έλεγχος. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. τροπολογία 4 υπέρ. Κατά κατά, αποχέσαι, ε, απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχέσαι, ε, εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχέσαι, εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ, κατά, αποχέσαι, εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ, κατά, αποχέσαι, εγκρίνεται. Τροπολογία 9 πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχέσαι, έλεγχος. Τέλος. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Yes, yes. We will do it again. We try again. Εντάξει, ωραία. Να το ξανακάνουμε ηλεκτρονικά την ψηφοφορία. Για το πρώτο τμήμα. Τροπολογία 9, πρώτο τμήμα, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται, ναι. Τώρα το δεύτερο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 12 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 13 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Τελική ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ για αυτές τις τροπολογίες. Η Επόμενη ψηφοφορία. Αφορά την δημοσιονομική διαδικασία και τον προπολογισμό. Η συγκέντρια είναι η κυρία Μπάρμπαρα Ματέρα. Φαμ 1 υπέρ. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείτε. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Θα ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας προφορίας. Απορρίπτεται. ΦΑΜ 2 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείτε. ΦΑΜ 3 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείτε. ΦΑΜ 4 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείτε. ΦΑΜ 5. Εδώ έχουμε 5 τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά το τρίτο τμήμα. Πέρας φοφορίας. Υιοθετείται. Τέταρτο τμήμα. Υπέρ κατά, εποχές απορρίπτεται. Πέμπτο τμήμα υπέρ, κατά, εποχές Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για να την ελέγξουμε. Πέρας προφορίας. Υιοθετείτε. Φάμε 6. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές υιοθετείται. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές ελέγχουμε. Ψηφίζουμε τώρα, ηλεκτρονικά. Τελειώνει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τέταρτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείτε. Πέμπτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε το πέμπτο τμήμα. Πέρα ψηφοφορίας. Υιοθετείτε. Φάμε 7 υπέρ. Κατά. αποχές Υιοθετείτε. ΦΑΜ 8. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείτε. ΦΑΜ 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείτε. ΦΑΜ 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείτε. ΦΑΜ 11. Υπέρ κατά εποχές υιοθετείτε, ΦΑΜ 12 υπέρ κατά εποχές υιοθετείτε, ΦΑΜ 13 πρώτο τμήμα υπέρ κατά εποχές υιοθετείται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά εποχές υιοθετείτε, Τρίτο τμήμα υπέρ κατά εποχές υιοθετείτε. ΦΑΜ 14 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές Υιοθετείτε. Το δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Πέραση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. Συγχαρητήρια για την εισηγήτρια. next point on the agenda. Το επόμενο σημείο είναι το 9 στη Μέση Διάταξη, η αποστολή στην Πολωνία. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, η έκθεση της αποστολή θεωρείται υιοθετηθήσα. 4 Σεπτεμβρίου, το απόγευμα θα κάνουμε την επόμενη μας συνεδρίαση. Δεν έχουμε κανένα άλλο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Σας εύχομαι και σε εσά και στις οικογένειές σας καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές. Ραντεβού το Σεπτέμβρη για τους κοινούς νητούς, εκτός από τους συντονιστές οι οποίοι θα πρέπει να παραμείνουν, γιατί σε λίγα λεπτά έχουμε τη συνάντηση των συντονιστών. Ευχαριστώ.